Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε την σύνοδο, την απογευματινή συνεδρίασή μας. Τα χθεσινά πρακτικά και τα εθετημένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Ε, υπάρχουν κάποια σχόλια. Έχετε επιφυλάξεις όσον αφορά αυτά που ανέφερα. Δεν βλέπω να υπάρχουν, οπότε θεωρούνται τα πρακτικά εγκεκριμένα. Πάμε στην ημερήσια διάταξή μας. Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επιτρέπουμε μία ώρα περίπου για αυτές τις συζητήσεις. Πρώτα σημείο, η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του blogger Σατάρ Μπεχέστη. Πρώτα απ' όλα, Ρωμίβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ιράν, στο Ιράν συνεχώς επιδεινώνεται. Πολλές περιπτώσεις βασανιστερίων, κακομεταχείρισης, αμελίες και θανάτους στο Ιράν έχουν καταγραφεί στον φυλακισμένους. Ο Μπεχέστη που ήταν 30 χρονών blogger συνελήφθη στις 30 Οκτωβρίου